Να αρχίσουμε κυρίες και κύριοι. Ήρθαν όλοι. I'm sorry that uh, we've uh, moved around from room to room. Συγγνώμη που περιφερόμεθα από αίθουσα σε αίθουσα, αλλά τι να κάνουμε. Πάντως αυτή είναι ωραία αίθουσα αυτή. Βλέπουμε και φυσικό φως, τον ήλιο α, έξω και πολύ χαιρόμαστε που ξαναβλέπουμε τον Μάριο Μόντι εδώ τρίτη, τέταρτη φορά. Πότε είναι από τότε που αρχίσατε αυτή τη σημαντική αποστολή, είχατε έρθει το Δεκέμβριο. Μια μεγάλη ανταλλαγή απόψεων για, μια, την έκθεση Μπρέτς που ήταν σημαντική και ακρογωνίως λίθος για τη δική μας την έκθεση γιατί τότε ε, είχαμε πει σοβαρά πράγματα που βρήκαν το δρόμο τους και στην έκθεση οπότε ήταν ένα ορόσημο. Παρακολουθούσαμε από κοντά την έκθεση. Είμαστε ευχαριστημένοι από το ξεκάθαρο και ειλικρινή τρόπο θα έλεγα με τον οποίο σκιαγραφίσατε κάποια προκλήσεις σε σχέση με τη νέα όθηση στην εσωτερική αγορά. Αυτό ήταν κομμάτι της, προσ... που προσωπικά είχατε αναλάβει. Εμείς ε, σας συγχαρήκαμε και για τη δουλειά σας και χάρη στον εισηγητή και μέσα από τον εισηγητή, από την κυρία Λούκας, και από τότε που εγκρίθηκε η έκθεση Louis Γκρέτς, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση του τύπου στο Στρασβούργο. Και βέβαια δεν ήταν τόσο διέδειξε τεράστιο ενδιαφέρον ο τύπος, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρευρισκόμενη. Αλλά και η κυρία Γκέμπχαρτ ε, και εγώ είδαμε τον Επίτροπο Μπαρνιέ και άλλους, τον Επίτροπο Ντάλι. Και ήταν και πολύ σημαντική αυτή η ε, επαφή Κοινοβουλίου Κομισιών για το σημαντικό θέμα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπουμε σήμερα το απόγευμα για να μας πείτε τι, τι, ποιας έτυχε η έκθεσή σας. Ποια είναι τα πιο προβληματικά ζητήματα που αποτελούν προκλήσεις ε, στους συνομιλητές σας. Τι προτάσεις γίνονται, αυτό ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει, είμαστε φιλόδοξη επιτροπή και μας ενδιαφέρει να μας πείτε και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, ποια είναι τα συμπεράσματα, τι συνέχεια θα δοθεί. Έχετε τον λόγο για να μας πείτε τις ιδέες σας και οι συνάδελφοι φαντάζομαι θα έχουν και κάποια ειδικά θέματα να σας θέσουν. Καλώς ήρθατε και με χαρά σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που είμαι τακτικός επισκέπτης και φιλοξενούμενος της Επιτροπής αυτής. Άλλωστε, εκτιμώ ιδιαίτερα τον κινητήριο ρόλο της Επιτροπής αυτής του Προέδρου της Μάλκολμ Χάρμπορ και του εισήγητη ε, Κρέγκ και τα άλλα θεσμικά όργανα την ίδια γνώμη έχουν, είμαι βέβαιος. Μου ζητήσατε κύριε Πρόεδρε να πω δύο λόγια για τα μετά της έκθεσης, γιατί η έκθεση Κρέγ. έπαιξε ρόλο κύριο σε σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία για τη νέα όθηση της εσωτερικής αγοράς, της ενιαίας αγοράς. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το εύρος, πλάτος, βάθος, ποικιλία του ενδιαφέροντος, όπως φάνηκε από τις διάφορες απαντήσεις, αντιδράσεις, η Κομισιόν πριν είναι κυρίως ε, το θεσμικό όργανο που ανέθεσε την έκθεση χάρη στην πρωτοβουλία του Πρόεδρου Μπαρόζο, ο οποίος Πρόεδρος Μπαρόζο με κάλεσε στη συνάντηση των Επιτρόπων στις 20 Ιουλίου, οπότε θα πάω για να παρουσιάσω θέματα, να συζητήσω και με εκείνον και με τους Επιτρόπους τη συνέχεια στο θέμα. Εν τω μεταξύ θα γίνουν διμερείς ε, συναντήσεις με τον Επίτροπο Μπαρνιέ κυρίως, αλλά και άλλους Επιτρόπους. Με χαρά μπορώ να πω ότι πολλοί Επίτροποι και οι υπηρεσίες τους άρχισαν να ενσωματώνουν τις αναλύσεις και συστάσεις της έκθεσης στις συνεχιζόμενες πολιτικές τους πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα έχετε ενημερωθεί ικανοποιητικά σχετικά με τις προθέσεις και τα πρώτα βήματα του Επιτρόπου Μπαρνιέ, οπότε εκείνος και όχι εγώ θα σας ενημερώσει. Αλλά εγώ έχω ενθαρρυνθεί πάρα πολύ από τις αντιδράσεις του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αυτή ειδικότερα υπήρξε και εξακολουθεί να είναι το βασικό σημείο αναφοράς για, αυτή, για αυτό το τομέα της πολιτικής, αλλά και αυτό είναι καλό νομίζω στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης υπέρ της οποίας στάσεται και η έκθεση Λούις Γκρέις και άλλες επιτροπές επίσης έδειξαν ενδιαφέρον στην Επιτροπή Απασχόληση, στην Επιστροπή Κοινωνικών Επιποθέσεων υπάρχει ενδιαφέρον για τη συζήτηση της έκθεσης. Και οι πολιτικές ομάδες επίσης δείχνουν ενδιαφέρον. Πολλές με κάλεσαν σε συναντήσεις για να συζητήσουμε την έκθεση και τη συνέχιση που θα της δοθεί. Το Συμβούλιο, μαζί σας κύριε Πρόεδρε, πήγαμε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, το Μάιο ήτανε, μάλιστα το Μάιο ήταν, ναι. Και η εντύπωσή μου είναι ότι αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για να μετρήσω με το βαθμό του ενδιαφέροντος και της αντιδράσης στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Όπως ξέρετε βέβαια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτησε την έκθεση και την πρόθεση της Κομισιόν να ε, δώσει συνέχεια σε αυτήν βράχη πρόθεσμα Και για να συμπληρώσω τις πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προσεκλήθη από τον πρόεδρο της ΕΕ να συζητήσω μαζί του και την το εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να συζητήσω λοιπόν την έκθεση και την προσέγγιση στην ενιαία αγορά και την Οικονομική Ένωση. Αυτό θα το κάνω σε 7 Ιουλίου στη Φραγκφούρτη. Οι εμπλεκόμενοι επίσης παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις εκδηλώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον. Να το Business Europe έχει το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό της ε, Συμβούλιο Σύνοδο Κορυφής τον Ιούλιο, 5 Ιουλίου και ασχολήθηκαν, ασχολούνται πολύ με αυτό το θέμα. Έχω επίσης επαφές με τα συνδικάτα, την Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα και πολλούς άλλους εμπλεκομένους και ενδιαφερομένους. Τώρα, τι μου λένε όλοι αυτοί. Νομίζω ότι η συνεργασία κατάφερε να ξαναβάλει στον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης την ενιαία αγορά, πράγμα που δεν συνέβαινε πριν από ένα χρόνο Και βλέπω όμως δύο μεγάλες προκλήσεις εδώ. Η μία είναι οι μεγάλες προσπάθειες που θεωρώ ότι ακόμη χρειάζονται για να πιστεί η κοινή γνώμη και οι πολιτικές ηγεσίε για τον κύριο ρόλο της ενιαίας αγοράς σε σχέση με τα δύο πιο σημαντικά θέματα σήμερα, την κρίση του ευρώ και την δημοσιονομική κρίση πολλών κρατών μελών. Αυτά τα δύο γεγονότα, όπως όλοι ξέρουμε, έχουν κάπως ε, υποβαθμίσει τη σημασία της ενίας αγοράς, αλλά οι πιο νυφάλιοι παρατηρητές βλέπουν όλο και καθαρότερα ότι ένας θεμελιώδης λόγος για την κρίση της Ευρωζώνης είναι στην πραγματικότητα η έλλειψη μιας οικονομικής ένωσης ε, στην Ευρωζώνη. Στη συνδιάσκεψη σήμερα ο Επίτροπος Φρανκ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του λέγοντας αυτά που έχουμε πει τόσες φορές εδώ εμείς ότι θα πρέπει να προσέξουμε πιο πολύ το ε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το, την Οικονομική Ένωση, που είναι ουσιαστικά η ενιαία αγορά. Και θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα την σύνδεση μεταξύ ενιαίας αγοράς και οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Γιατί λόγω της δημοσιονομικής κρίσης είναι αδύνατο να προέλθουν τα ενάβσματα για την μεγέθυνση από τον προϋπολογισμό. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν τα, η όθηση αυτή να έρθει από το σκέλος της προσφοράς μέσα από ένα μεγάλο άλμα στην δομή διάρθρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, δηλαδή την ενιαία αγορά. Χρειάζονται να γίνουν πολλά ακόμα λοιπόν και στα πλαίσια της διαμόρφωσης της κοινή γνώμης για τα δύο αυτά και το δεύτερο και τελευταίο σημείο είναι μια ανησυχία ουσιαστικά. Όπως γνωρίζετε στη προσέγγιση μου και τη νέα στρατηγική που παρουσιάστηκε στην Κομισιόν υπάρχει αντίληψη περί ενός πακέτου. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί περισσότερο ή λιγότερο για ένα ε, ή το άλλο στοιχείο του πακέτου, αλλά είμαι πεπισμένος ότι χρειάζεται μια ευρεία ε, προσέγγιση πακέτου. Χωρίς πακέτο μπορεί να υπάρχουν πολλές καλές προθέσεις, αλλά τα παραδοτέα, όπως λέμε, θα είναι πενιχρά τα τελικά αποτελέσματα και τα περισσότερα μονομένα μέτρα που όλοι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά για να δοθεί όθηση στην ενιαία αγορά προσκρούν σε αντιστάσεις εδώ και εκεί και νομίζω ότι είναι δύσκολο να ε, υπερκεράσουμε αυτές τις αντιστάσεις. Θα είναι δε αδύνατον απολύτως να ξεπεράσουμε τις αντιστάσεις εκτός και αν δημιουργηθεί ένα πακέτο όπου ο καθένας θα βρίσκει κάτι το καλό. Μπορεί να είναι δύσκολο να τα καταπιούν όλα, αλλά να έχουν και κάτι που να τους αρέσει, κάτι που να αρέσει σε ένα κράτος μέλος ή σε ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Αυτό για μένα είναι ένα θέμα κλειδί. Αλλά αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι εάν θέλουμε να επιτελέσουμε σημαντική πρόοδο, νομίζω ότι τα ανώτερα ηγετικά κλιμάκια θα πρέπει να δεσμευτούν προσωπικά. Δηλαδή, μιλάω αφενός για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι αισιόδοξο εδώ, γιατί στο κάτω-κάτω ανέλαβε δράση εντοπίζοντας την ενιαία αγορά ως ε, βασική πολιτική προτεραιότητα για την, ε, στα πλαίσια της δεύτερης θητείας του και από την άλλη και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει επίσης να το νιώσει αυτό ως μια προτεραιότητα. Γιατί μόνο έτσι θα είναι πιστεύω δυνατόν οι δράσεις των επιμέρους τομεακών συμβουλίων, ανταγωνιστικότητας κοινωνικών υποθέσεων, εκοφήν κλπ. θα μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερη συνοχή στη δράση τους. Από αυτή την άποψη, και αυτή είναι η τελευταία μου λέξη κυρία Πρόεδρε, η ιδέα ενός νομοθετικού fast track που μας αρέσει και στους δύο, μια ταχεία διαδικασία, νομίζω ότι είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση. Με δύο λόγια, Κατά τη γνώμη μου η κεντρική δέσμευση δεν θα πρέπει να είναι τόσο η λεπτομερή συζήτηση της τάδε ή της δίνα πρότασης, αλλά μάλλον πώς από κοινού μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο της δημιουργίας, ίσως αυτό έγινε ήδη, αλλά διατήρησης της ε, πολιτικής σημασίας του θέματος αυτού παρά την πληκτική ε, δήθεν η επιφανειακά τεχνοκρατική και γκρίζα μορφή που μπορεί καμιά φορά να παρουσιάζεται μπροστά μας, την, όχι τόσο ελκυστική. Ευχαριστώ πολύ Μάριο για την ενδιαφέρουσα αυτή ανασκόπηση ήθελα να δώσω το λόγο στο Λουί Γκρέσ να απαντήσει πρώτος. Αυτό θα ήταν το πιο ενδεδειγμένο, αλλά επιτρέψτε μου κάνα δύο σχόλια προηγουμένως. Ε, μας ε, ε, ενθάρρυνε η αντίδραση στη δουλειά μας, γιατί ο Επίτροπος Μπαρνιέθ βλέπει τώρα με αυτόν τον τρόπο την σημασία της ενιαίας αγοράς, γιατί το μήνυμα από εμά είναι ότι η ενιαία αγορά αφορά καταναλωτές, πολίτες, γιατί ε, και εσείς στην εκθεσή σας είπατε ότι πρέπει οι ψηφοφόροι να στηρίξουν την ενιαία αγορά, οι καταναλωτές, οι πολίτες, γιατί έτσι θα μπορέσει να εξελιχθεί και να βελτιωθεί και η διακυβέρνηση. Και υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες εκεί για το πώς θα γίνει αυτό, όπως ας πούμε να έχουμε ένα κατάλογο των 20 βασικών παραπώνων που έχουν οι πολίτες από την ε, ενιαία αγορά. Αυτό μάλιστα γίνεται τώρα, διερευνάται. Οπότε ήταν μια άμεση αντίδραση αυτή, ούτως ώστε το πολιτικό κέντρο βάρους να βγει από τα τεχνοκρατικά θέματα και να αποκτήσει ευρύτερο χαρακτήρα. Και ο Λουί ε, που συγκέντρωσε τις 180 ψήφους υπέρ ήταν πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην το πρόσεξαν πολύ αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούν ε, όλες οι πολιτικές ομάδες. Καλό θα ήταν λοιπόν ο Λουί Κρέξ, ο οποίος είναι εισηγητής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, να πάρει πρώτο το λόγο για να απαντήσει. Και μετά ο κύριος Σφάμπ, Γκέπχαρ, Γουζόη, Ρούλαρ, οι σκληρά εργαζόμενοι συντονιστές μας. Λοιπόν, ας βάλουμε μπρο και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μπορεί να, ακούμε, να τους ακούμε τρεις-τρεις και να απαντάτε, να δούμε πώς θα γίνει. Μετά κρατσα Βιλτ Κορέντε Κάμπος, ε, κυρία Ράπτη, ε, κυρία Βάιλερ επίσης και πολλοί άλλοι. Αλλά ξέρω ότι θα μείνετε μέχρι τις τέσσερις. Ε, οι συνάδελφοι όμως ε, θέλουν να παραμείνουν τελευταία. Μετά αρχίζει και το ποδόσφαιρο. We are Συμφωνούμε, κύριε Μόντι, όταν λέτε ότι η ενιαία αγορά είναι λιγότερο δημοφιλής από ποτέ. Επίσης συμφωνούμε ότι η ενία αγορά θα πρέπει για τους πολίτες, για τους ε, καταναλωτές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υλοποιήσει τους στόχους, αν θέλουμε μια υψηλά ανταγωνιστική οικονομία. Αλλά πιστεύω ότι τα μηνύματα της Επιτροπής είναι μεικτά. Απ' τη μία, ο Επίτροπος Μπαρνιέ είναι πολύ ενεργητικός, ε, θετικός, γεμάτος ζήλο και προωθεί συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για την ανανέωση αναζωγόνηση της ε, ενίας αγοράς, ενώ ο πρόεδρος Μπαρόζο, ο οποίος λέει ότι είναι ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας η ενία αγορά, δεν θέτει την ενία αγορά στις βασικές πρωτοβουλίες στρατηγικής 2020. Είναι δυνατόν, παρότι είναι ακόμα δυνατόν να πούμε ότι η τρίτη πρόκλησή σας που αναφέρατε, ε, με κάποια αυταρέσκεια και θεωρείται ότι η ενιαία αγορά είναι παλιά ε, προτεραιότητα, όχι σημερινή, όχι σύγχρονη. Ε, υπάρχει αυτή η αντίληψη σε ορισμένου αξιωματούχους κομισιών. Ο κύριος Φάμπα. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο εισηγητής μας για το κείμενο που μας έδωσε ο κύριος Μόντι. Κύριε Μόντι, είπατε ότι πρέπει να συνεισφέρουμε ε, ώστε να πείσουμε την κοινή γνώμη για τα πλεονεκτήματα της ενιαία αγοράς. Και στη δημοσιονομική κρίση, στην οικονομική κρίση, είδαμε ότι πολλοί πολίτες θεωρούν ε, ότι υπάρχουν ωφέλη από την εσωτερική αγορά, μιλάω για τη χώρα μου βέβαια, αλλά θεωρούν ότι είναι αυτονόητα τα πλεονεκτήματα, ενώ οι υποχρεώσεις, ε, αλλά ότι οι δυνατότητες που ανοίγονται δεν είναι τόσο ελκυστικές. Θα πρέπει λοιπόν να επηρεάσουμε θετικά την κοινή γνώμη και ε, σε σχέση με την ανησυχία που εκφράσατε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί πακέτο η πρόταση, εδώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι δύσκολο να πούμε ότι θα δεχτούμε συνολικά το πακέτο σας ως βάση για την πολιτική μας δουλειά, γιατί παρόλο που σε πολλούς τομείς συμπίπτουν οι απόψεις μας, παρόλα αυτά βλέπουμε και άλλες δυνατότητες παρέκκλησης ή υπέρβασης των προτάσεών σας. Με ενδιαφέρει να μου πείτε ποια είναι τα σημαντικότερα θεωρείτε μέτρα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν σημαντικά τμήματα αυτού του πακέτου. Ε, βέβαια είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά ίσως μπορείτε να μας πείτε τα σημαντικότερα ε, συστατικά στοιχεία του πακέτου όπως το φαντάζεστε. Ευχαριστώ. η Εύλιν Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που μας βοηθάει πολύ. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να στηριχθούμε σε δύο βασικές αρχές όπως τις επεξεργαστήκατε στην, ε, στο κείμενό σας κύριε καθηγητά Μόντι ε, η συνολική λύση όπως είπατε η οποία μπορεί να ε, παρουσιαστεί και να προβληθεί και να ψηφιστεί με έναν ενιαίο και όχι αποσπασματικό τρόπο. Και αυτό το συνδέω και με την έννοια του πολιτικού οράματος, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε στην πολιτική, σε, αυτό, σε αυτή την πολιτική. Και αν ε, αποφασίσουμε τι όραμα επιδιώκουμε, τότε θα είναι πιο εύκολο να συνεννοηθούμε και με τους πολίτες και όχι να τους πούμε αυτό είναι πάρτε το. Ε, ένα άλλο θέμα που απορρέει και από την έκθεση Λουί Κρέχ για τον κατάλογο των 20 ε, βασικών παραπώνων. Ξέρω ότι αυτό το επεξεργάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να κάνουμε πια ένα βήμα ακόμα και να πούμε εντάξει, δεχόμα, γινόμαστε παραλήπτες των παραπώνων. Αυτό Αυτά τα παράπονα όμως εκφράζουν ανάγκες, έτσι δεν είναι και πρέπει εκεί να δώσουμε απαντήσεις. Όχι δηλαδή με τρόπο αρνητικό να σχολιάσουμε τα παράπονα των πολιτών, αλλά να δούμε τι θετικές ενέργειες μπορούν να συνδεθούν με αυτά για να λυθούν τα προβλήματα. Αυτό είναι που πρέπει να το ε, προωθήσουμε στο προσκήνιο πολύ περισσότερο. Και αν είναι και αυτό αυτός και δικό σας στόχος, τότε εγώ και η ομάδα μου είμαστε 100% στο πλευρό σας. Τώρα, λέω να δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Μόντι να απαντήσει για να μην έχουμε πολλές ερωτήσεις μαζί, αλλά κυρία Κοράτσα Μπίλτα πήγεται να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Ε, μπορούν και άλλοι συντονιστές να θέσουν τα σχόλιά τους τώρα και μετά ο κύριος Μόντι να σχολιάσει τις πρώτες ερωτήσεις και μετά να δώσω το λόγο στο, στην κυρία Ρούλερ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, έχω αεροπλάνο, πρέπει να φύγω 4 παρατέταρτο. Ε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μόντι. Είναι πολύ επίκαιρη η έκθεσή σας, γιατί η οικονομική ανάκαμψη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σημαίνει ότι πρέπει να θέσουμε εκ νέου της, την ενιαία αγορά στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα εστιάσουμε στην πραγματική οικονομία. Το ερώτημά μου, πώς θα τα καταφέρουμε και πώς θα εφαρμόσουμε, πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, ποιες είναι οι απόψεις σας για να λάβουμε υπόψη μας τις πολιτικές ανησυχίες και τις ανησυχίες των πολιτών. Και μάλιστα θέλω να στραφώ και προς την Κομισιόν εδώ και να καλέσω την Κομισιόν να δώσει συνέχεια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πάρα αυτά συμπεριλαμβάνοντας την πρόταση για την πράξη της ανίας αγοράς στις συστάσεις του κύριου Μόντι. Κύριε Μόντι, ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκεκριμένα βήματα από εδώ και πέρα για να εφαρμόσουμε τις συστάσεις σας. Τι πρέπει να κάνουμε, πολύ συγκεκριμένα. Ο κύριος Μόντι, κύριε Γκρέχ, σας συγχαίρω ακόμα μια φορά για την έκθεσή σου, για την έκθεσή σας και υπάρχουν ε, σημεία σύγκληση μεταξύ του δικού μου κειμένου και του δικού σας. Καταλαβαίνω ότι στην ε, στρατηγική για την, ε, για την Ευρώπη του 2020 δεν υπάρχει η ενιαία αγορά ως βασική προτεραιότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικού ενδιαφέροντος δεν νομίζω ότι είναι αυτό ο λόγος. Νομίζω ότι απλώς η ενιαία αγορά ε, δίνει αυτό το πολιτικό, πολιτική όθηση, αν θέλετε, στη στρατηγική 2020. Δεν θέλω να τη δω έτσι απομονωμένα και χαίρομαι για την ε, έντονη ζέση του Επιτρόπου Μπαγνιέ, που είναι και αρμόδιος, για την, αρμόδιος επίτροπος για την ενιαία αγορά. Αυτό που προτείνω στην έκθεσή μου είναι κάτι το οποίο πηγαίνει ακόμη πιο πέρα από αυτά που είπαν οι επίτροποι σε, αυτό σε αυτήν την ομάδα των επιτρόπων ε, της οποίας προεδρεύει ο κύριος Μπαρνιέ. να σας διαβάσω τέσσερις γραμμές από το κείμενό μου. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει ηγετικό ρόλο για να εξασφαλίσει ένα συνολικό όραμα. Μια ομάδα επιτρόπων που θα έχουν όλες τις αρμοδιότητες για την οικονομική ολοκλήρωση υπό την ε, προεδρία του Προέδρου ή του Επιτρόπου ε, Ενίας Αγοράς και Υπηρεσιών σε περίπτωση που απουσιάζει ο πρόεδρος μπορεί να είναι το κατάλληλο σώμα για τη διατύπωση πολιτικών προτάσεων. Αυτό που δημιουργήθηκε τώρα είναι μία ομάδα όντως επιτρόπων υπό την Προεδρία του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, αλλά φυσικά αν παραστεί ο πρόεδρος, αν παρίσταται ο πρόεδρος, θα προεδρεύει αυτός αυτής της ομάδας. Είναι περίπου αυτό που πρότεινα και εγώ. Πέρα όμως από τις διατυπώσεις και τα τυπικά, Μια και έζησα τη ζωή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 10 χρόνια, καταλαβαίνω ότι αυτό που είναι σημαντικό, ο κάθε επίτροπος να αισθάνεται ότι έχει τα κίνητρα για να αναπτύξει το δικό του τομέα, τις δικές του πολιτικές, τις αρμοδιο... στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με... στα πλαίσια των βασικών στόχων της ενίας αγοράς και της οικονομικής ολοκλήρωσης. Ίσως αυτό θα ήταν πιο εύκολο να επιτευχθεί αν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παίζει ένα ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί μπορεί οι επίτροποι να μην έχουν τόση ζέση και τόση όρεξη να συνεισφέρουν αν ε, αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό την ηγεσία Ενό άλλου συναδέλφου και όχι του Προέδρου. Ε, είναι αυτό ένα μικρό πρόβλημα. Αλλά ξέρω ότι ο πρόεδρο εν ενδιαφέρεται. Και φαντάζομαι ότι θα βρεθούν οι κατάλληλε λύσει και η σωστή οργάνωση. προ τον κύριο Σβάμπ. Σέβομαι και συμφωνώ με το σχόλιο σας. Ότι μια προσέγγιση τύπου πακέτου δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε υπέρ όλων. Θυμάμαι ε, στα ηλίσια στο ίδιο παλάτι που ήταν παρούσα και η κυρία Γκέπχαρτ και θυμάμαι και τα μέλη της Επιτροπής Αταλή που, θέλαν να, που είχαν ετοιμάσει μάλλον την γαλλική έκθεση για την ε, γαλλική οικονομία. Ο πρόεδρος Ζάκα θυμάστε ότι ήταν πολύ τολμηρός, είπε στον πρόεδρο και όλα αυτά τα μετέδει η τηλεόραση. Πρόεδρε, έχουμε 316 προτάσεις εδώ. Ή θα πρέπει να τις δεχτείτε όλες ή να τις απορρίψετε όλες. Γιατί υπάρχει απόλυτη λογική αλληλουχία μεταξύ τους. Αυτά το 2008, έτσι, τον Ιανουάριο του 2008. Ε, και ο πρόεδρος Μπορείτε να φανταστείτε πώς αντέδρασε σε αυτόν τον ε, επιμέρους διάλογο με τον Ζακατέλη. Σωστό είναι λοιπόν κύριε Σφάμπ αυτό που είπατε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα επιμέρους σημεία. Αλλά μην ξεχνάμε και το όλο. Επιμένω ότι πρέπει να υπάρχει πακέτο. Και αυτό ε, συνδέεται με την προηγούμενη απάντηση που δώσα. Όποια και να είναι τα μέτρα, τα καλύτερότερα. Και αν αφορούν αποκλειστικά τις, ε, τις αρμοδιότητες της ενίας αγοράς, που είναι ούτως ή άλλως ε, ευρείες, δεν θα αρκούν παρόλα αυτά. Δεν αρκούν από μόνο τους. Γιατί υπάρχουν κοινωνικές ε, πτυχές, γιατί υπάρχουν βιομηχανικές πτυχές, βιομηχανικής πολιτικής δηλαδή, εμπορικής, ε, εμπορικές πολιτικές και εξωτερικών σχέσεων, ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, φορολογικά στοιχεία, φορολογικές πολιτικές. Επομένως, χρειάζεται το πακέτο ούτω ώστε να υπάρξει τελικά γενική συμφωνία. Μια προκαταρτική απόφαση θα ληφθεί Καταρχά επί του ιδίου του πακέτου, το χρειαζόμαστε ή όχι. Και από εκεί και πέρα, σε μια δεύτερη φάση, πρέπει να συζητήσουμε τα επιμέρους στοιχεία. Αλλά σε δεύτερη φάση, κυρία Γκέπχαρτ. Μου αρέσει ο θετικός τρόπος με τον οποίο βλέπετε αυτά τα 20 πιο συνήθη παράπονα που τα αντιμετωπίζετε ως μια προσπάθεια διερεύνησης. Ποια είναι, ποιες είναι οι μεγαλύτερες φιλοδοξίες, αν θέλετε, μελήματα που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα των πολιτών. Δεν είναι αυτοτιμωρία, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ε, δεν είναι αυτομαστίγωμα, είναι προσήλωση στο, στα ενδιαφέροντα και στις ανησυχίες των πολιτών. Είναι πιο επικοδομητική δηλαδή η προσέγγισή σας. Πιο έξυπνη θα έλεγα κιόλας. Κυρία Κοράτσα Μπίλτα. Αρχικά σκέφτηκα να σας μιλήσω Ιταλικά, αλλά μιλήσατε Αγγλικά. Δυστυχώ δεν μπορώ να σας μιλήσω Σουηδικά πάντω, όπως και να έχει. Σας ευχαριστώ για τις, ε, ε, τα σχόλιά σα ε, για τα θετικά που είπατε. Σημαντικό αυτό που αναφέρατε για την ανάγκη να δοθεί έτσι πολιτική σημασία και να προωθηθεί, αν θέλετε, η πολιτική διάσταση της ενίας αγοράς. Οπουδήποτε και αν πηγαίνει κανείς, σε οποιαδήποτε φόρουμ για να συζητήσει ευρωπαϊκά θέματα, Και μάλιστα εσείς όταν πηγαίνετε, οπουδήποτε και αν πηγαίνετε, σε οποιαδήποτε βήματα, ε, πάντα προωθείτε αυτή την θεώρηση ε, συνεχίστε το. Και αυτό που είπατε για την ανάπτυξη, για τη δυσκολία να βρεθούν άλλες πηγές ανάπτυξης στην Ευρώπη, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει για να προωθήσουμε πιο δραστήρια την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Μας δώσατε πολλές ιδέες. Και άλλες, περισσότερες ιδέες. Αλλά αυτό που είπατε ότι η αγορά, ότι τροφοδοτεί έτσι την πολιτική συζήτηση, την πολιτική όθηση αν θέλετε, για τα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 είναι ενδιαφέρον. Ε, νομίζω ότι η Κομισιόν ε, η ίδια, και η δική μας επιτροπή θέλουμε να παίξει αυτό το ρόλο έτσι, της ατμομηχανής αν θέλετε. Πουσόι Ρούλε, Ρούλερ, Πουσόι Κάμπος, Τριανταφυλλίδης, αυτοί τέσσερις. Μπουζόη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μου απαντήσετε Ιταλικά. Ξέρετε ότι εμεί ε, αγαπάμε πάρα πολύ τα Ιταλικά, οπότε ευχαρίστω να σα ακούσω να μου απαντάτε Ιταλικά. Συγχαρητήρια για τι διαβουλεύσει αυτέ που έχετε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε και πολύ θα ήθελα να είχαμε και περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε το πακέτο σας. Τώρα ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε την εφαρμογή του πακέτου. Εγώ πιστεύω ότι θέλουμε και χρειαζόμαστε ένα φιλόδοξο πακέτο. Και χρειαζόμαστε πολύ σχηρά μέτρα σε πολλούς τομείς. Ένα πακέτο λοιπόν με πολλά μέτρα είναι μια καλή ιδέα. Υπάρχουν όμως μερικά προβλήματα που δεν είναι εύκολο να λύσουμε. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα και ίσως μπορούμε να βρούμε κάποια λύση. Για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου πολίτες που πάνε σε άλλη χώρα και θέλουν να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα ή να ανοίξουν λογαριασμό στη χώρα αυτή, αντιμετωπίζουν πολύ περίεργες καταστάσεις. Γιατί σε ορισμένες χώρες δεν μπορείς να νοικιάσεις διαμέρισμα δεν έχεις τραπεζικό λογαριασμό και δεν μπορείς να ανοίξεις τραπεζικό λογαριασμό αν δεν δώσεις διεύθυνση. Καταλαβαίνετε πόσο παράλογη είναι αυτή η κατάσταση. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς μπορούμε να λύσουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κατά τα άλλα η αμοιβαία αναγνώριση αυθεντικών πράξεων, μια κάρτα για ελεύθερη κυκλοφορία, ίσως είναι κάτι που μπορούμε πιο εύκολα να θέσουμε σε εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Ρούλα, ευχαριστώ και εγώ για τη δουλειά σας. Καλό είναι που τονίζετε την ε, διατηρησιμότητα, νέες προκλήσεις από την οικολογική, όχι μόνο τη δημοσιονομική κρίση και καλό είναι να το δούμε όλα αυτά ως πακέτο. Έχω την εντύπωση όμως ότι η Κομισιόν δεν το βλέπει αναγκαστικά ως τέτοιο και φοβάμαι ότι ενδεχομένως θα επικρατήσουν μεμονωμένες εξατομικευμένες απόψεις. Καλό θα ήταν να μπορούμε να συζητήσουμε για τα μέτρα και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί θα πρέπει να πείσουμε και αυτούς που είναι οι ενάντι στο εγχείρημα της ε, ενιαία αγορά και αυτοί που είναι επιφυλακτικοί και αυτοί που θα είναι οι υπέρμαχοι, όλοι να συμμετέχουν σε, σε ένα κοινό εγχείρημα. Καλό είναι αυτό και σωστό, αλλά αν δούμε που ασκείται η περισσότερη κριτική σήμερα στην εσωτερική αγορά συνδέεται με την ε, δημοσιονομική κρίση. Γιατί πολλοί λένε ότι έγιναν λίγα πράγματα, ότι άνοιξαν οι αγορές, αλλά δεν ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των καταναλωτών, ούτε οι μηχανισμοί ελέγχου. Και το θέμα είναι τώρα, θα τα καταφέρουμε. Βλέποντας τη διάθεση στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ περιορισμένες οι ε, προθέσεις και τα οράματα. Μου φαίνεται ότι παρά είστε απεσιόδοξοι. Θα περιμένουμε να δούμε. Ο κ. Δεκάμπος. Ευχαριστώ. Όπως περνάει ο καιρός, έχω την εντύπωση στην έκθεση Μόντι βλέπουμε το πρώτο σημάδι αισιοδοξία των τελευταίων καιρών. Είναι μια σφαιρική έκθεση που κερδίζει υποστηρικτέ, που εμπνέει τον κόσμο και δημιουργεί ενθουσιασμό. Είναι ένα από τα ελάχιστα θετικά σημάδια που είχαμε τον τελευταίο καιρό με την οικονομική αυτή κρίση. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που διαπιστώνω την ε, προσέγγισή σας. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά πρέπει να αυξήσουμε την κατανάλωση. Και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι και αυτήν ακριβώ τη δουλειά για να ενθαρρύνουν την κατανάλωση και όχι να κάνουμε το αντίθετο όπω γίνεται. Προσπαθούμε ορισμένοι, ας πούμε, ο Ομπάμα προσπαθεί να αναβάλει την ε, κατανάλωση. Όμως εγώ νομίζω ότι το αντίθετο πρέπει να κάνουμε και δεν ξέρω πώς μπορούμε να αυξήσουμε την κατανάλωση. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε να κάνουμε αυτά που προτείνετε στην έκθεσή σας κύριε Μόντι. Είναι μια δουλειά που πρέπει να την κάνουμε ώστε η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να αυξηθεί. Γιατί αν λιμνάζουμε, ε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει. Κύριε Μόντι, τώρα εσείς μιλάτε πολύ προσεκτικά, διαλέγετε τα λόγια σας. Αλλιώς περιγράφετε την συνεισφορά του Πρόεδρου της ε, Επιτροπής για τα επόμενα βήματα και αλλιώς περιγράφεται ε, τα πράγματα από πλευρά του Συμβουλίου, του Πρόεδρου του Συμβουλίου. Μήπως πρέπει ακόμα να πείσουμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, μήπως πρέπει, πρέπει να τον πείσουμε να εμπλεχθεί και να στηρίξει και αυτός την έκθεσή σας. Σίγουρα εσεί μπορείτε καλύτερα να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε από ότι εγώ. Αλλά έχουμε τρεις μεγάλες ευκαιρίε εδώ. για να προχωρήσουμε με την ενία αγορά. Την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών πρώτα απ' όλα, όπου πρέπει να αξιολογήσουμε και την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η οδηγία αυτή για τις υπηρεσίες δεν ήταν τόσο θετική και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν, οι υπηρεσίες. Και το τρίτο είναι η ελεύθερη διακίνηση των επαγγελματιών. Ούτε και εδώ είχαμε μεγάλη επιτυχία. Έχουμε λοιπόν δουλειά μπροστά μας. Καλά θα κάνουμε να ξεκινήσουμε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε κύριε Μόντι να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους για τα καλά σας λόγια. Κύριε Μπουζόη, το δίλημα που θέτεται, το τρομερό αυτό δίλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη για να εγκατασταθούν αλλού, ε, φοβάμαι ναι ότι οδηγεί σε ένα διέξοδο. Όντως είναι ένας φαύλος κύκλος. Ε, για να έχεις ε, λογαριασμό χρειάζεται διεύθυνση και για να έχει σπίτι χρειάζεται λογαριασμό τραπεζικό. Πραγματικά είναι τρελό. Δεν είμαι δυστυχώς σε θέση να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση αυτή τη στιγμή, μια λύση. Αλλά θα περιλαμβάνετε. Α, υπάρχει ήδη στα 20 σημεία. Στα 20 παράπονα των πολιτών. γιατί εδώ η πίεση του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου πρέπει να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Διότι δεν πρέπει να είναι τόσο δύσκολο πια για να λυθεί κάτι τέτοιο. Και καταλαβαίνετε τι ζημιά κάνει στην ενιαία αγορά. Περιπτώσεις σαν κι αυτήν. Κύριε εσείς λέτε ότι στην έκθεση αναφέρουμε πολλά για τη βιωσιμότητα. Δύο φορές αναφέρεται ο όρος sustainability στην έκθεση. Η μία φορά είναι επειδή μιλάμε για την ενιαία αγορά, την πράσινη ανάπτυξη, το περιβάλλον, αλλά αν σκεφτούμε καλά όλο αυτό το εγχείρημα έχει να κάνει με το να έχουμε μια ολοκληρωμένη αλλά και βιώσιμη αγορά. Γιατί τι διαπιστώσαμε, το ξέρετε κι εσείς από την καθημερινή σας πολιτική εμπειρία επιτόπου. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των αγορών σταδιακά διαβρώνεται, υπονομεύεται και καταστρέφεται. Προσπαθούμε λοιπόν στην έκθεση να διατυπώσουμε, να εκφράσουμε αυτές ακριβώς τις ανησυχίες ώστε να μην υπάρχουν πια εμπόδια στη συνέχιση της ολοκλήρωσης των αγορών μας. Αυτή λοιπόν η έννοια της βιωσιμότητας είναι όντως μια πολύ δυνατή έννοια. Μας βοηθάει να ε, φτιάξουμε τις πολιτικές μας για την ολοκλήρωση των αγορών. Και είδαμε το πρόβλημα που είχαμε και με την οικονομική κρίση, με την πρόσβαση στις δυσιονομικές αγορές. Γι' αυτό και μιλάω για μία κόποση όσον αφορά την ολοκλήρωση. Αλλά θα έλεγα ότι πρόκειται ίσως και για κόπωση των αγορών. Και καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο έχει αυτό στους καταναλωτές. Πάντως δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος όσο εσείς για το μέλλον, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτά που κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να τα ανταπεξέλθουν, να φροντίσουν να υπάρχει ένα εποπτικό πακέτο, για παράδειγμα, η θέση που υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προωθηθεί, να συσταθεί παρετέρω. Και εμείς είμαστε πολύ κοντά στο Κοινοβούλιο, περισσότερο από ό,τι στο Συμβούλιο. Κύριε Κάμπος. Ναι, πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση. Γιατί πράγματι είναι κάτι που πάει χέρι-χέρι με την ανάπτυξη της αγοράς. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση όμως σε μια περίοδο όπου ε, θέλουμε να περιοριστούν τα ελλείμματα, τα δημοσιονομικά. Και έτσι ερχόμαστε σε κάτι που συζητήσαμε και νωρίτερα. Πώς να πετύχουμε περισσότερη ανάπτυξη. μέσω μιας ε, μεγαλύτερης ολοκλήρωσης στις ε, αγορές. Βλέπετε, θα σας δώσω μια ιδέα. Η Γερμανία έχει να παίξει ένα ρόλο κλειδί, αναμφίβολα, όπως πιστεύουν πολλοί Ευρωπαίοι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχει και πολύ νόημα να κάνουμε αυτό που κάνουν πολλοί. Δηλαδή, να πιέσουμε τη Γερμανία προκειμένου να ξοδεύει περισσότερα για να στηρίξει την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι η Γερμανία δεν αυθυγραμμίζεται έτσι με τη δικιά της ηθική φιλοσοφία θα έλεγα. Δεν λέω ότι η κατανάλωση είναι κακό, εκείνη σχεδόν αυτό νομίζει. Αν λοιπόν ε, τώρα χρησιμοποιηθεί και για το δημοσιονομικό έλλειμμα, μήπως καλύτερα να πιέσουμε τη Γερμανία να μην είναι και ενησιακή, αλλά να είναι γερμανική. Για να πάμε πίσω στο Λούδι Γκέραρτ. για την οικονομική κοινωνική οικονομία της αγοράς, οικονομία και κοινωνία που διέπουν την αγορά. Ξέρετε τη σχολή του Φράγκμπουργκ και την κοινωνική οικονομία. Χάρη στη Γερμανία έχουμε τον ανταγωνισμό στη συνθήκη και η Γερμανία μετά την επανένωση έγινε λιγότερο ενθουσιώδης για όλα αυτά από ό,τι ήταν αρχικά. Εγώ πάντως πιστεύω και πολλοί Γερμανοί οικονομολόγοι το πιστεύουν επίσης ότι εάν η Γερμανία άνοιγε περισσότερο, ελευθέρωνε περισσότερο το τομέα των δικών της δημοσίων υπηρεσιών, αυτό θα ήταν κάτι που θα πήγαινε προς την κατεύθυνση περισσότερη αγορά στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Με το βάρος που έχει η Γερμανία θα μπορούσε να δείξει το δρόμο και αντί να εμποδίζει την ολοκλήρωση. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δούμε μια συμμαχία ανάμεσα στη γερμανική κυβέρνηση και την ευρετανική κυβέρνηση. Κάτι που δεν το περιμέναμε. Και μαζί να ε, μπουν σε μια νέα περίοδο όθησης της οικονομίας στην Ευρώπη. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε πολύ σοβαρά. Κύριε Κάμπος, η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε τότε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση. Όχι όμως μέσω κινήτρων στον προπολογισμό. Οι Γερμανοί δεν θα δεχόντουσαν κάτι τέτοιο. Τέλος, μας δίνεται τρεις ε, βάσεις δικαιώματα των καταναλωτών, οδηγία για τις υπηρεσίες και ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών. Είναι τρία πράγματα, μεταξύ άλλων, που όντως πρέπει να δοκιμαστούν. Αναφερθήκατε επίσης στον πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Εγώ ήδη πριν από μερικούς μήνες είπα ότι κατά τη γνώμη μου είναι αποφασιστική σημασία ο ρόλος του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Στην έκθεσή μου όμως λέω κάτι και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Το εξή. Τώρα που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μέσα από το ρόλο του μόνιμου Πρόεδρου μπορεί να προσφέρει περισσότερη συνέχεια στην ε, οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθούσε αν είχαμε ένα υψηλού επίπεδου κατευθυντήρια γραμμή για τη συνεισφορά του Συμβουλίου σε αυτό το στοιχείο κλειδί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης που είναι η ενιαία αγορά. Εννοείται ότι το δικαίωμα πρωτοβουλίας και επιβολής παραμένει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως όλη η διαδικασία για να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στην ενιαία αγορά είναι κάτι που μπορεί να πετύχει εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όχι οποιαδήποτε, όχι οποιαδήποτε συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φροντίσει να δώσει στον πρόεδρό του την εντολή να προσφέρει συνέχεια στο θέμα αυτό, σε στενή συνεργασία βέβαια με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, είδαμε 30 και παραπάνω χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταλήξει όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Ανεπιτυχώς. Και αυτό έχει να κάνει και με ανεπαρκή ηγεσία στο Συμβούλιο. Γιατί αυτό δεν είναι πρόβλημα της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, είναι του Συμβουλίου η ηγεσία του Συμβουλίου, ίσως και εξαιτία του συστήματος περιτροπής προεδριών, δεν τα κατάφερε. Τώρα έχουμε ένα μόνιμο πρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, θέματα τα οποία είναι ζητικής, ζωτικής σημασίας για την εσωτερική αγορά και που κολλάνε στις διάφορες ομάδες του Συμβουλίου, θα πρέπει να πάνε στην Προεδρία του Συμβουλίου η οποία θα φροντίσει να τους δώσει κάποια συνέχεια, να προσφέρει κάποια συνέχεια από την οποία όλοι έχουμε να αποφεληθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές. Κύριε Μόντι, όχι ό,τι λέτε εσείς ότι δεν ε, σας θες το ύψος, όχι εμείς πιστεύουμε πως ναι, τα χαιρόμαστε όλα αυτά και σας διαβεβαιώνω ότι Υπάρχουν επαφές μεταξύ Λονδίνου και Βερολίνου. Μην ανησυχείτε, υπάρχουν αυτές οι επαφές. Και περιμένουμε φυσικά να δούμε τα αποτελέσματα. Το άλλο είναι ότι εγώ έγραψα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ζήτησα να έρθει στην Επιτροπή μας. Γιατί όντως μετά την παρουσίαση για την στρατηγική του 2020 θα βοηθούσε έτσι κι αλλιώς, με στην ελπίδα ζούμε. η κυρία Ράπτη, η κυρία Βάιλερ και ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Οι κυρίες πρώτα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας άλλος συνάδελφος που θέλει το λόγο. Για την, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την έκθεση που μας παρουσιάσατε. Σας άκουσα με πολύ προσοχή και εδώ και χτες στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, τα λέτε πολύ ωραία και θα έλεγα ότι φραστικά αγγίζεται όλα τα ζητήματα με χειρουργικό τρόπο. Ε, αγγίζεται οικονομικά ζητήματα, αλλά και βαθύτατα πολιτικά ζητήματα. Μας έχετε δώσει ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά βάζετε ε, έναν όρο που ε, με μία λέξη το είπατε μία φορά. Βάζετε το θέμα της ταχύτητας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο όπως μας είπατε αν δεν χρησιμοποιηθεί γρήγορα, τότε το εργαλείο αυτό θα μείνει άχρηστο. Δεν θα μπορέσει να δώσει τα αποτελέσματα για τα οποία σχεδιάστηκε. Και θέλω να σας ρωτήσω ε, με ποιο τρόπο νομίζετε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ταχύτητα στη δράση, όταν προηγουμένως μας περιγράψατε, για παράδειγμα, πως εάν προεδρεύσει της Επιτροπής των Επιτρόπων ο κύριος Μπαρνιέ μπορεί να μην έχουμε τόσο γρήγορα αποτελέσματα όσο αν προείδρευε ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής γιατί οι υπόλοιποι επίτροποι δεν θα δέχονται ευχάριστα μια άλλη προεδρία. Αυτό τουλάχιστον ε, έφτασε στα αυτιά μου. Και η ερώτησή μου είναι αυτή, το γρήγορα πώς εξασφαλίζεται. Thank uh, Mrs. Weiler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μη φοβάστε, δεν θα αρχίσω το γερμανικό ζήτημα, να το αναλύω. Αλλά επανέρχομαι σε ένα θέμα καθηγητά Μόντι. Ε, κάνατε μια μικρή κριτική και συμφωνώ ε, στη Γερμανία και είπατε ότι σε ορισμένους τομείς δεν ανοίγει την αγορά η Γερμανία. Καταλαβαίνουμε τι εννοείται. Ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Ένα. Ξέρετε όμως και γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ δεν είμαι υπέρ του ανοίγματο μόνο μέσα από τη σκοπιά της εσωτερικής αγοράς, αλλά και διότι είναι δικαίωμα των εργαζομένων η ελεύθερη διακίνηση, να μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν πού θα δουλέψουν στην Ευρώπη. Εκεί έχει ένα πρόβλημα η Γερμανία, το οποίο όμως έχει να κάνει και με τους μισθούς dumping. Είναι θα ήταν εξαιρετικό να προτείνατε στην Κομισιόν και ένα νόμο, μια οδηγία κατά των ε, αμοιβών dumping, ελάχιστων μισθών dumping, Ξέρω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις εδώ σε ό,τι αφορά το ύψος. Επίσης, σε άλλους τομείς η Ευρώπη έχει εργατικού δικαίου διατάξεις κατά των διακρίσεων ωραιότατες, τις οποίες εμείς ευχαρίστως ε, εφαρμόσαμε. Ίσως μπορεί και εδώ να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πολλοί Γερμανοί εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα έρθει ξένο εργατικό δυναμικό που θα ρίξει ή θα δουλεύει με μισθούς ένα τρίτο χαμηλότερους και έτσι ο κοινωνικός ιστός της χώρας ε, θα ε, ζημιώσει. Επίσης καλό θα ήταν στη ρησομιλία σας να εξηγήσετε περισσότερο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσα από εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα, πανεπιστήμια, ΑΕΗ ε, γιατί υπάρχουν ελάχιστοι που τάσσονται υπέρ των περικοπών στην ε, παιδεία. Αυτό δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ένωσης. Δεν πρέπει να γίνει δεκτό. Γιατί ε, θα βραχικυκλώσουν έτσι όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και τα πιο πετυχημένα σκανδιναβικά κράτη. Πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση, έρευνα. Βλέπουμε τι κάνουν οι ασιατικές χώρες. Και καλό θα ήταν και στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσο σημαντική είναι η έρευνα και η παιδεία και να μην έρθει στο κεφάλι κάποιας χώρας μέλους να ε, βάλει μπρος περικοπές στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ κύριε Στερενταφυλίδης. Θα παρακαλούσα τον προφέσορ Μόντι να ενδιατρύψει ο λίγον στο λέξη package μήπως αυτό παραπέμπει σε ένα μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης και το ερωτώ αυτό παρότι στην έκθεση γίνεται διαχωρισμός των προσεγγίσεων με βάση το οικονομικό σύστημα και τη γεωγραφική τοποθεσία των χωρών. Και αυτό είναι ενδεικτικό ότι στην ενιαία αγορά συμμετέχουν σήμερα οικονομίες με διαφορετικές προτεραιότητες. Συνεπώς, η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την εσωτερική αγορά θα πρέπει να συνδυάσει τις αξίες και τις αρχές του κάθε μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης. Έχω την εντύπωση ότι η επιμονή στην εφαρμογή ενός προτύπου για όλα τα κράτη, ανεξαρτήτως εθνικών ιδιαιτεροτήτων, θα δημιουργεί πάντοτε προβλήματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρότσμαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Είναι εξαιρετική η έκθεσή σας γιατί στις αναλύσεις σας διαπιστώνετε ότι πρέπει να γίνει. Και κάνετε και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, πράγμα σπάνιο για εκθέσεις. Δεν λέτε γενικά, γενικόλογα τι πρέπει να γίνει, αλλά βάζετε στη, έναν οδικό χάρτη και λέτε αυτά και αυτά πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρουμε, για παράδειγμα, από τον κύριο Μπαρνιέ, ότι ε, έχει αντίκτυπο η έκθεσή σας στην τωρινή δουλειά. Η εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντική για το είδος ανάπτυξης της Ευρώπης, γιατί είναι τεράστια η δυναμική της, τα λέτε, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τόσα άλλα. Και επίσης ε, και τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους εκεί που έχουν αρμοδιότητα, δικαιοδοσία, στον κοινωνικό τομέα, στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να αναλάβουν δράση, γιατί το συνταγματικό δικαστήριο, για παράδειγμα, το συνταγματικό δικαστήριο δεν ε, δίνει πολλά περιθώρια. Μία μικρή ερώτηση. Λέτε για την ελεύθερη διακίνηση που είναι θαυμάσια προϋπόθεση για τους εργαζομένους. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Μπουζόη, ε, έτσι ανοίγει γενικότερα η αγορά. Αλλά τι θα πρέπει να έχει η κάρτα ας πούμε ελεύθερης διακίνησης για κοινωνική ασφάλιση, εγκατάσταση κλπ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πρόβλημα με αυτούς που ε, τάσσονται υπέρ της προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να τα γράφει αυτά η κάρτα. Για την εσωτερική αγορά θα λειτουργούσε ρότατα μια τέτοια κάρτα και για τον εργαζόμενο, για να μπορέσει να δείξει ότι έχει άδεια εργασία, ότι συντρέχουν όλε οι προποθέσει για την ελεύθερη διακίνηση. Το free movement card είναι εξαιρετικό πράγμα. Αλλά φοβάμαι ότι θα έρθουν αυτοί που προστατεύουν πάντα τα ιδιωτικά δεδομένα και θα μας κάνουν δυσκολίες. Thank you very much indeed. Um... Ευχαριστώ να ασκήσω και εγώ το προνόμιο του Προέδρου κάνοντας ένα-δύο σχόλια και ρωτώντας ένα-δύο πράγματα. Υπάρχουν διάφορες συστάσεις προς το Κοινοβούλιο, τις οποίες εξετάζουμε, ιδίω στο κεφάλαιο που μιλάτε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου, λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα εξασφαλίσει μια πιο ενιαία θεώρηση και όραμα στην ενιαία αγορά, εμπλέκοντας περισσότερες ε, επιτροπές. Αν έχετε κάποιες ιδέες για το πώς το πετύχουμε, ε, μπορείτε να μας πείτε, α πούμε, οι υπόλοιπε επιτροπές πώς ε, υποδέχτηκαν την έκθεσή σας. Κάτι άλλο, πιο συγκεκριμένο, γιατί οι συντονιστές της Επιτροπής αυτή τη στιγμή εξετάζουν τι μελλοντικέ πολιτικέ πρωτοβουλίε μα για να προχωρήσουμε τα πράγματα. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σημαντική ατζέντα ε, που αναφέρεται στο κεφάλαιο 4. Ε, πώς θα υλοποιήσουμε μια ισχυρή αγορά. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από την πολιτική μας υποστήριξη. Παραδείγματο χάρη, πώς θα δημιουργήσει τις δυνατότητες αυτές η Επιτροπή πώς θα τις προωθήσει με τα γραφεία αυτά και με το Solvit. Ε, διάφορα πράγματα λέτε εκεί. Θα μπορούσατε να, μας, ε, να μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να υπάρξει εφαρμογή. Πώς μπορούμε ας πούμε, να υλοποιήσουμε αυτές τις ιδέες. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις ερωτήσεις και σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά που με προσκαλέσατε στην Επιτροπή σας. Προς την κυρία Ράπτη. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ταχύτητα. Πφ, δύσκολο ερώτημα. Ακούγοντας και το πρώτο σχόλιο του Προέδρου, δηλαδή τη προς το, αυτό που είπε για τη συστάση μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Διερωτώ με, μήπως εσείς, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας όλος ιδιαίτερος θα μπορούσατε να βοηθήσετε περισσότερο πιέζοντας, οθώντας τους πάντες να περάσουν σε μια ανώτερη ταχύτητα. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι παρέκβαση, Πρόεδρε, συγχωρέστε με. Θα μπορούσατε λοιπόν να το κάνετε πιέζοντας τα άλλα δύο θεσμικά όργανα για να δημιουργήσουν έτσι, μια ετήσια, πώς να την πω, γιορτή, μια ευκαιρία, ας πούμε, όπου θα δίδονται ομιλίες, θα γίνονται ομιλίες για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, την κατάσταση της, πώς προχωράει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε οικονομικό επίπεδο. Υψηλού επίπεδου συνάντηση, πολιτικού επίπεδου, με πολιτική διάσταση, μια πολιτική στιγμή, αν θέλετε, όπου αποτυπώνουμε και αποτιμούμε το τι έχει γίνει που θα μπορούσε να αντισταθμίσει, αν θέλετε, την ε, εξόχως κατακαιρματισμένη φύση αυτών των συζητήσεων. Νομίζω ότι θα ήταν μια ευκαιρία όπου κάθε θεσμικό όργανο, σε αυτά τα πλαίσια αυτής της ε, ετήσιας, αν θέλετε, ομιλίας, μια και εσείς έχετε τον, ε, την απαλλαγή, έτσι, στον τομέα του προπολογισμού. Κάτι αντίστοιχο έχω στο μυαλό μου, κάτι αντίστοιχο με την απαλλαγή να έχουμε μια ευκαιρία όπου θα λέμε τι έκανε ο καθένας, πόσο αποτελεσματικά, πόσο βοήθησε στην οικονομική ολοκλήρωση, πόσο συνεισέφερε. Κάθε λεπτό οι αγορές και η κοινή γνώμη δίνουν τεράστια προσοχή σε κάτι που είναι πολύ λιγότερο σημαντικό, το ενιαίο νόμισμα τελικά. Και δεν δίνουν καμία προσοχή στην ενιαία αγορά. Όλη η εστίαση πάει στο ενιαίο νόμισμα. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο, σχηματικά τα λέω. Αλλά εσείς είστε αυτοί και κυρίω η Επιτροπή σας που είναι η καρδιά αυτής προσπάθειας που μπορείτε να απαιτήσετε μια από κοινού περιοδική αποτίμηση της κατάστασης. Και μιλάμε για ένα θέμα που αφορά και τους 27, έτσι, όχι τους 16. Αυτό, κυρία Ράπτη, νομίζω θα μπορούσε να αυξήσει λίγο την ταχύτητα. Κυρία Βάιλερ. Καθώς μιλούσατε, εγώ σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν πόσο αναγκαίο είναι αυτό το πακέτο που προωθώ. Γιατί αναφέρονται κάποια παραδείγματα που ήταν τέλεια και που δημιουργούν, που εγείρουν κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικά ερωτήματα. Αν δεν επιλύσουμε αυτά τα κοινωνικά ζητήματα, δεν θα υπάρξει πρόοδος στην εσωτερική αγορά και στην ελεύθερη κυκλοφορία κτλ. κτλ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπάρξει οδηγία της Επιτροπής εναντίον των dumping στους μισθούς. Θα έλεγα μάλλον καλύτερα αυτό που είπε η κυρία Ράπτη. Αυτή τη χειρουργική ας πούμε επέμβαση, πιο εστιασμένη. Στην έκθεσή μου μιλάω για δύο ε, σημεία του συστήματος που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων. Λαβάλ, έκθεση Λαβάλ κτλ. Μετά τις επαφές που είχαμε την Business Europe, μπορούμε να διερευνήσουμε κάποιες ατραπούς. Ο Επίτροπος το εξετάζει. Και κάτι άλλο που είναι ευρύτερο, είναι ο συντονισμός των φόρων, φορολογικός συντονισμός. Αντί να επιβάλλουμε από τις Βρυξέλλες μια εναρμονισμένη κοινωνική πολιτική, ας επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να μπορούν να συνεχίζουν τις δικές τους κοινωνικές πολιτικές, χωρίς να αισθάνονται ότι τους περιορίζουν ε, ασφικτικά με τον φορολογικό ανταγωνισμό και τους αφαιρούν τις αρμοδιότητες τις φορολογικές ε, και με αυτόν τον τρόπο διαβρώνουν και τη φορολογική τους βάση και χάνουν και τα φορολογικά τους, αν θέλετε, δικαιώματα. Κύριε Τρενταφυλλίδη, για την ε, οικονομική διακυβέρνηση, ε, ομογένεια, οικονομικά μοντέλα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει μια λύση, μια πανάκια, κάτι που είναι καλό για όλα. Και αυτό που με ελκύει διανοητικά που με ήλκησε στη δουλειά που έκανα τουλάχιστον και ελπίζω να μην χαθεί. Παραδείγμα, σας, σας παρακαλώ παρα, πιο συγκεκριμένα στο follow-up της Κομισιόν ε, να μην τις επιτρέψετε να δημιουργήσει με βάση την έκθεσή μου ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, να προσθέσουμε αυτό, εκείνο και το άλλο, άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Επανέρχομαι. Αυτό που βρίσκω ελκυστικό είναι η εξή ιδέα. Να εμπλακούν χώρε οι οποίε έχουν διαφορετική οικονομική φιλοσοφία. Η οικονομία τη κοινωνική αγορά, της υπηρετική Ευρώπη, τους Αγγλοσάξονες, τα νέα κρατημέλη. Όλοι αυτοί μαζί να βρούνε αντισταθμίσει που ελπίζω να έχω περιγράψει. ούτω ώστε να αρθούν οι δικαιολογίε, οι φόβοι, για να βάζουν τροχοπέδι στην ενιαία αγορά. Δεν μπορώ ότι πρέπει να επιβάλλουμε εκ των άνω ένα εναρμονισμένο μοντέλο. Θα πρέπει, κυρία Ράπτη, χειρουργικά, όπως είπατε, να πάμε να δούμε πού υπάρχει, σε ποιο μοντέλο υπάρχουν τραυματισμοί. Και αν δεν ε, χειρουργηθούν αυτοί, θα υπάρξει μια μόνιμη απόλυτη υποστροφή προς την ανάπτυξη της ε, εσωτερικής αγοράς. Κύριε Πρόεδρε, σας απάντησα στην αρχή της παρέμβασής μου. Ε, για τις συστάσεις που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησα. Ναι, αυτή η παρέκβαση που κανά ε, για αυτή την ετήσια ομιλία κτλ. Αλλά είχατε και μια δεύτερη ερώτηση, κάπου μου ξέφυγε. Αφορούσε τις συστάσεις σας στο γενικό κεφάλαιο για την υλοποίηση μιας στεναρή μιας αγοράς. Θα κάνω και εγώ μια παρέκβαση. Έτσι, σχέδια. Μήπω θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τους συντονιστές ε, να μας επιτρέψουν μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία, όπου εκεί θα λάβουμε υπόψη μα τι συστάσεις. Γιατί είναι μια δέσμη συστάσεων πραγματικά συνεκτική. Ε, έχετε διάφορες, μας δίνετε διάφορες ιδέες, ας πούμε το Solvit, ε, κάνετε διάφορες προτάσεις συγκεκριμένες. Απάντηση. Έχετε μια συνήθιστη ικανότητα να χρησιμοποιείτε αυτή την, αυτό το χαρτί των εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας. Φαντάζομαι λοιπόν, ε, όπως κάνατε και στο παρελθόν, ε, και τώρα θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε τους καταλληλότερους, τους εξυπνότερους ε, εισηγητές. Για Μάριο Μόντι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα είναι η τελευταία φορά, ελπίζουμε. Η έκθεσή σου αποτελεί για μιας μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία για να σε φωνάζουμε εδώ, αλλά κάθε ευκαιρία είναι καλή. Χαίρομαι λοιπόν για όσα μας είπες, ακόμα και εκτός θέματος, πάντα τα χαίρομαι αυτά. Όπως είπε και η κυρία Ράπτη, η χειρουργική σου προσέγγιση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άκουσα και αυτό που υπόθηκε επίσης για την πολιτική ενέργεια. Ε, λοιπόν, και εμείς πιστεύουμε, εδώ στην Επιτροπή μας, ότι εσείς μας προσφέρετε αυτή την πολιτική ενέργεια και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια μας. Τροφοδοτείτε με νεολικό. εντάξει, δεν ακούσαμε Ιταλικά, αλλά πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Και η Ιταλία χάσατε, χάσατε και την αρχή του μάτς που ξεκίνησε στις 4. Κυρίες και κύριοι, ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο με τον ε, καθηγητή Μόντι, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να υποφεληθούμε από την εμπειρία του. Και τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα. Έχουμε χρόνο. είναι ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε για την γνωμοδότησή μας, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, η οποία ετοιμάζει με συγκίτα την κυρία Νίμπλερ την επί της ουσίας έκθεση για τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων. Εμείς έχουμε την κυρία Βάιλερ από τη δικιά μας την πλευρά, που είναι η συγκίτρια για την γνωμοδότησή μας. Για να δω πόσους σκιώδες έχω. Ο κύριος Βαντεκάμ δεν είναι εδώ. Α, έρχεται. Ο κύριος Κρότσμαν είναι εδώ. Κύριε Ρούλε, όσο εδώ ήτανε. Δεν είσαστε. Είσαστε εδώ τώρα, αλλά θα έχετε κάποιον άλλον. Το σκιώδη σας περιμένετε. Θα έρθει φαντάζομαι. Εγώ είμαι σκιώδης από τη δικιά μου την πολιτική ομάδα. Ο κύριος Δεγιόγκ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Δαβίνη ούτε. Ο Ζων Βότσον είναι εδώ από το τμήμα της Γενικής Γραμματείας που είναι η Διεύθυνση ΓΑΜΑ. Καλώς. Έχουμε ένα έγγραφο εργασίας της κυρίας Νίμπλερ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Βάιλερ για να μας εισαγάγει στο θέμα και να μας εξηγήσει την προσέγγιση της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνουμε εξαντλητική συζήτηση σήμερα, γιατί είμαστε στην αρχή της συζήτησης. Η κυρία Νίμπλερ συνέταξε ένα ενδιαφέρον έγγραφο, αλλά από ό,τι γνωρίζω για την Επιτροπή τη νομική, όχι τη δική μας. Εμείς θα διαφοροποιήσουμε λίγο την έμφαση σε σχέση με την νομική επιτροπή. Αλλά είναι πολύ καλό που συμμετέχουμε κι εμείς. Επίσης νομίζω ότι είναι σωστό, είναι σωστή η βασική απόφαση το συνολικό πακέτο να το δούμε και στα πλαίσια του Better Regulation, του Κρήτων Νομοθετήν. Ε, και ε, θα συμπεριλάβουμε και επιτυχίες του Λούι Γκρέχ για την εσωτερική αγορά, δηλαδή να δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα τα θέματα επίσης. Τώρα, καταρχήν τι περιμένουμε από μια νέα διαμόρφωση των κειμένων. Θέλουμε να συμμετέχουμε ως κοινοβούλιο. Μέχρι τώρα τι έχει γίνει. Έχουν, υπάρχουν εκτιμήσεις επιπτώσεων εδώ και κάποια χρόνια και λεβέ και στα κράτη-μέλη γίνονται εκτιμήσεις επιπτώσεων που όλες όμως ε, σκοπό έχουν να δουν τι στοιχίζει, ποιο είναι το κόστος μιας νομοθεσίας. Σωστό είναι αυτό, αλλά εμείς δεν θα περιοριστούμε εκεί, θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Όχι μόνο τις δαπάνες, το τι στοιχίζει ένα ε, νομοσχέδιο, αλλά θα δούμε και άλλα πράγματα. Διάβασα με ενδιαφέρον το κείμενο της κυρίας Νίμπλερ που μεταξύ άλλων λέει ότι έχει νόημα να δούμε κάποια στιγμή τις best practices, βέλτιστες πρακτικές που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ε, τα όρια μας ποια συστήματα υπάρχουν στη Σκανδιναβία, Σουηδία και την Ολλανδία αναφέρει η κυρία Νίμπλερ. Μου φαίνεται ότι θα έρθει η Βέλγος ή Ολλανδός σκιώδης από τους συντηρητικού. Έτσι ακούω. Θα, ε, είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί η Ολλανδία είναι η μόνη χώρα μέλος που για την περαιτέρω συνέχιση των εργασιών ε, υποχρεούται να δημοσιεύει όλες τις πληροφορίες. Ενδιαφέρει και η Αμερική, αλλά ας δούμε πρώτα τι, έξω από την πόρτα μας. Αν υπάρχει κάτι στη Σουηδία και την Ολλανδία που να μπορούμε εμείς να το μιμηθούμε, σίγουρα θα είναι καλό. Τώρα, οι βασικές αρχές που κατέγραψε η κυρία Νίμπλερ με βρίσκουν σύμφωνοι καταρχήν ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων μπορεί να είναι μόνο βοήθημα για την πολιτική λήψη αποφάσεων, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη διαδικασία, ούτε επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Βέβαια το ερώτημα είναι από πού θα αρχίσουμε πριν από την νομοθεσία μετά, τη θέσπιση της νομοθεσίας ως κοινοβούλιο, θα πρέπει μετά να κάνουμε κάποια εκτίμηση επιπτώσεων και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, ευτυχώς το θέλαμε από καιρό. Είμαστε πια υποχρεωμένοι να κάνουμε τέτοια εκτίμηση επιπτώσεων και θα δούμε πού θα την βάλουμε, πώς θα τη συνδέσουμε και πώς θα ενταχθεί και το Κοινοβούλιο στις διαδικασίες αυτές. Η κυρία Νίμπλερ λέει ακόμη ότι η εκτίμηση επιπτώσεων δεν πρέπει να οδηγούν σε καθυστερήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να γίνεται και παράλληλα η εκτίμηση αυτή, ούτε θα πρέπει να γίνονται μηχανιστικά για να αποφεύγουμε ανεπιθύμητες ε, ε, νομικές διατάξεις. Γιατί το, το είδαμε και αυτό κάποιες φορές. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι αρκετά ισχυρό, όμως ούτω ώστε να αντέξει σε αυτούς τους πειρασμούς. Και μου φαίνεται ότι και η Κομισιόν είναι το ίδιο ισχυρή. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό για μας στις μελλοντικές οδηγίες, πρωτοβουλίες ε, της Κομισιόν, κανονισμούς, πρωτοβουλίες για να το πω γενικά, να λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα προστασίας των καταναλωτών που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα, γιατί η εκτίμηση επιπτώσεων κόστους δεν είναι ε, εξαντλητική, ούτε λαμβάνει υπόψη όλες τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία, έτσι για να το πω ουδέτερα, αλλαγές. Δεν θα ήταν άσχημο νομίζω να κάνουμε κάτι που εν μέρη κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή ένα SME τεστ, Βέβαια, τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια σε, δραστηριοποιούνται ήδη σε πολλούς τομείς που δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε κι εμείς. Πάντως εγώ δεν έχω προ... υπάρχουσα άποψη, ήδη δηλαδή διαμορφωμένη άποψη για το ποιος θα κάνει το... τη μελέτη επιπτώσεων θα είναι εσωτερικός, θα είναι εξωτερικός. Οι εξωτερικοί δυσκολότερα ελέγχονται η διαδικασία είναι λιγότερο διαφανής από ότι αν γίνει εσωτερική η δουλειά αυτή και δεν είμαι και βέβαιος ε, αν είναι και πιο οικονομική από το να το κάνουμε εμείς μόνοι μας. Πάντως, εγώ θα ενημερωθώ για τις απόψεις των άλλων, γιατί είμαστε στην αρχή. Δεν έγινε ε, συζήτηση στην ομάδα μου για αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό πάντως στο μέλλον πέρα από τα οικονομικά ζητήματα να εξετάζονται τα οικολογικά, τα κοινωνικά, τα κοινωνικά αυτά που αφορούν τους καταναλωτές. Αυτή είναι η άποψη της ομάδας μου και η δική μου προσωπικά και αν το καταφέρουμε σίγουρα θα έχουμε βελτιώσει το σημερινό status quo. Γιατί δεν αρχίζομαι από το μηδέν, ήδη, υπάρχει κάποια σημαντική εμπειρία συγκεντρωμένη, υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν best practices και έτσι με την ησυχία μας θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να διαμορφώσουμε μια άποψη σχετικά με την καλύτερη λύση ενός προβλήματος που όλοι έχουμε εντοπίσει και που όλοι θέλουμε να ε, λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Um, suffering from an absence of shadows this afternoon, but Mr. is uh, loyal to the ends. And... Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κρότζεν και μετά θα δούμε ποιος άλλος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Ε, θα κάνουμε πριν από τα νομοθετήματα τις εκτιμήσεις επιπτώσεων για να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν, αλλά και μετά να δούμε δηλαδή αν αυτά που πιστεύαμε γίνανε. Επίσης στις εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει να σκεφτόμαστε συμβάλλουμε στην αύξηση της γραφειοκρατίας μήπως ποιες είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις, ποιες είναι οι επιπτώσεις της θέσης εργασίας. Πολύ σημαντικό αυτό θεωρώ για να δούμε αν με τις οδηγίες μας δημιουργούμε θέσεις εργασίας ή μήπως τις καταστρέφουμε καταστρέφουμε θέσεις εργασία βραχυπρόθεσμα, ε, αυξάνουμε ε, γενικά τις ευκαιρίες. Ε, επίσης, στο... το τεστ επικουρικότητας δεν θα το απέριπτα, γιατί υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. εμένα δεν θα με νοιάζει ποιος θα κάνει την εκτίμηση επιπτώσεων, αν θα το κάνει η Κομισιόν με το δικό της προσωπικό ή αν θα το αναθέσει σε τρίτους. Το σημαντικό είναι να γίνουν οι εκτιμήσεις με αντικειμενικά κριτήρια και να μην, είναι, να μην έχουν πολιτικά, πολιτικό χρωματισμό. Να μην αναθέσει κάποιος δηλαδή μια εκτίμηση επιπτώσεων και να είναι προδιαγεγραμμένο και το αποτέλεσμα. Όχι, να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Είναι καλό λοιπόν, εγώ θα Περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει. Θα συμβάλλουμε και εμείς επικοδομητικά. Ε, έχουμε αναφέρει κάποια σημαντικά για μας θέματα και θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας δείξει η κυρία Βάιλερ ως ε, πρώτο σχέδιο και μετά θα συνεχιστεί η συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ωραία. Όπως οι σκιώδες εισηγητές, έτσι και εγώ έχω κάποιε παρατηρήσει Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε μπροστά μας από τότε που ήρθα στο Κοινοβούλιο. Εγώ βέβαια θα κατευθυνθώ διαφορετικά. Διότι αυτό που εμένα με απασχολεί στην προσέγγιση της κυρίας Νίμπλερ είναι ακριβώς ο όρος ανεξάρτητο. Διότι σημαίνει ότι άμα έχουμε ανεξάρτητους θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Έτσι όπως το θέτει. Εγώ όμως δεν είμαι πεπισμένος καθόλου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μια ανεξάρτητη αξιολόγηση που να έρχεται κάποιος δηλαδή απ' έξω και να αξιολογεί τη δουλειά που έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Αν αυτό εννοεί με τον όρο ανεξάρτητη, δεν ξέρω. Εδώ πέρα πρόκειται σαν να διαχωρίζουμε τις ευθύνες, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό ως εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλει η κυρία Νίμπλερ, υποθέτω, είναι να υπάρχει αντικειμενικότητα. Δηλαδή οι αξιωματούχοι να έχουν μια αντικειμενική άποψη για τις θέσεις τους και τη δουλειά τους. Και γι' αυτό θέλει έναν ανεξάρτητο που θα εκτιμήσει αυτή την αντικειμενικότητα. Κάποιοι συνάδελφοι εδώ στο Κοινοβούλιο πιστεύουν ότι ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα πάει σε κάποιον άλλον για να το αξιολογήσει. Όχι, αυτό δεν θα ήταν σωστό κατά τη γνώμη μου, θα ήταν λάθος. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμείς εδώ δεν είναι μια καθαρά μηχανιστική προσέγγιση που να λέει ότι κάθε πρόταση θα εξετάζεται από την ανεξάρτητη αρχή και θα αναλύεται. Όχι. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς κυρία Βάιλερ, αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε ε, να κάνουμε τη δουλειά καλύτερα. Και ό,τι πολιτική προτείνεται πρέπει να γίνεται βάσει μιας πολύ προσεκτικής διαδικασίας όπου θα αναλύεται κάθε φορά και συστηματικά τις αναλλακτικέ λύσεις που έχετε για να δείτε και να τις συγκρίνετε με τους στόχους και μετά να αποφασίζετε ποια εναλλακτική λύση είναι καλύτερη. Και αυτό είναι μία εκτίμηση επιπτώσεων. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει. Είμαστε η μόνη επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου όλοι οι συντονιστέ και βουλευτέ βουλευτές συμφώνησαν πριν πάρουμε πρόταση για έλεγχο πρέπει να γίνεται εκτίμηση επιπτώσεων. Και εσεί, κυρία Βάιλερ που είσαστε και η συγγήτρια για τις πληρωμές ξέρετε ότι είσαστε οι πρώτοι στο Κοινοβούλιο που αναλαμβάνει κάτι τέτοιο. Θα συμφωνήσετε ότι όλη η συζήτηση που είχαμε για την εκτίμηση επιπτώσεων βοήθησε πάρα πολύ τους βουλευτές. Θυμόσαστε πόσοι πολλοί είμαστε, τι ανάλυση είχαμε και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ανάλυση για τις αναλλακτικέ λύσεις και μας εξήγησαν γιατί επέλεξαν κάποια πρόσθετα μέσα και αποφάσισαν να τα υποστηρίξουν. Ε, αυτό λοιπόν θέλουμε να γίνεται. Αλλά αυτή δεν είναι δουλειά που μπορείτε να αναφέσετε σε κάποιον εξωτερικό. Θέλουμε καλή νομοθεσία, θέλουμε καλή δουλειά. Η αξιωματική έχει της Επιτροπής που πιστεύω ότι κάνουν δουλειά υψηλής ποιότητας. Πρέπει να κάνουν και αυτό. Είναι μέρος της δουλειά τους. Και όντως πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να ξέρουμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές και να γίνεται συστηματικά αυτή η αξιολόγηση και να διατίθεται και σε μας. Είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και άνοιγμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το θέλουμε. βοηθάει στη χρηστή και κυβέρνηση. Αλλά δεν θέλετε αυτό να το αναθέσετε σε εξωτερικούς, σε outsiders. Θα το ξέρετε. Το σύνδρομο αυτό έχετε δουλέψει σε οργανώσεις. Αλλάζει η διαχείριση και τελικά αναθέτεται έξω σε κάποιον να εκτιμήσει τη δουλειά σας. Και τι κάνετε τότε, προσπαθείτε να μυθείτε, να εξηγήσετε τι καλή δουλειά κάνετε και μετά να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτεροι και από τους consultants. Αν αναθέσετε έξω την εκτίμηση επιπτώσεων, κατά τη γνώμη μου, θα καταλήξουμε σε χειρότερη νομοθεσία. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε. Από την άλλη μεριά, αν έχουμε αντικειμενική ανάλυση ποιότητας, που μπορεί να ελεγχθεί από εξωτερικούς, τότε εντάξει. Δεύτερον, πρέπει να καταρρύψουμε το επιχείρημα εκείνο που λέει μερικές φορές πρέπει να κάνουμε τα πράγματα τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε εκτίμηση επιπτώσεων. Μα κάθε καλά συνταγμένη πρόταση πρέπει να ακολουθεί διαδικασίες και λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν και την εκτίμηση επιπτώσεων. Αν δεν υπάρχει ο χρόνος, για εκτίμηση επιπτώσεων, ε, τότε δεν έχουμε και χρόνο να ε, μελετήσουμε και να εγκρίνουμε ή όχι την πρόταση. Διότι αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει προηγουμένω η σωστή ανάλυση, η αντικειμενική που πρέπει να γίνεται πριν καταλήξει σε πρόταση. Αυτό το επιχείρημα λοιπόν πρέπει να το καταρρύψουμε. Και ελπίζω ότι θα με υποστηρίξουν οι συνάδελφοι σε αυτό. Τέλος, όσον αφορά τα κριτήρια και την ανάλυση. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα θέματα που έχουμε μπροστά μας σήμερα και καλό είναι που το συζητάμε είναι ότι οι εξελίξεις όσον αφορά την εκτίμηση, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων δυσκολεύει και παγώνει την όλη συζήτηση. Η εκτίμηση επιπτώσεων δεν είναι μια και Πρέπει να έχει άμεση σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Άρα πρέπει να βλέπουμε τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή είναι μια πρώτη αξιολόγηση εκτίμηση επιπτώσεων, και άπαξ και έχουν γίνει επιλογές στη στρατηγική, μετά ακολουθεί η νομοθετική πρόταση. Και πιστεύω ότι ο τρόπος ε, με τον οποίο δουλεύει η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται. Δηλαδή τι κάνουμε. Ε, κάνουμε λίγο πολύ ότι κάνουμε και με τις εκθέσεις μας ιδίας πρωτοβουλίας. Επιλέγουμε τις στρατηγικές και μετά μιλάμε για τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας. Το επιχείρημά μου λοιπόν είναι εδώ ότι όσο περισσότερο χρόνο ε, ξοδέψετε για να κάνετε την ανάλυση σας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε όσον αφορά την νομοθετική πρόταση. Και δεν νομίζω ότι σας καθυστερεί αυτό τελικά. Γιατί αν το Κοινοβούλιο είναι πεπισμένο για τη στρατηγική, είναι πολύ πιο εύκολο να προχωρήσουμε στις λεπτομέρειες. Το είδαμε και σήμερα το πρωί. Εδώ στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε για τη δομή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Γιατί δεν πέρασε από αυτή τη διαδικασία. Ήταν μια φτωχή εκτίμηση επιπτώσεων για αυτή την πρόταση. Αν είχαν εκτιμηθεί η στρατηγική και είχε συζητηθεί στην προηγούμενη θητεία και είχαμε αποφασίσει την κατεύθυνση που θα παίρναμε, ελάχιστη εναρμόνιση, δομή της πρότασης κτλ, θα είχαμε τελειώσει με την νομοθετική διαδικασία τώρα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του γιατί δεν πρέπει να βιαζόμαστε στην ε, εκτίμηση επιπτώσεων. Δεν πρέπει να δεχτούμε ποτέ το επιχείρημα που λέει ότι «Μα δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε καιρό για εκτίμηση επιπτώσεων». Όχι, γιατί τότε πλήττεται τη διαφάνεια. Και δεν έχουμε αρκετά καλή ε, νομοθετική πρόταση. Από πλευρά τη Επιτροπή μας, θυμηθείτε τι μας είπε ο καθηγητής Μόντι, όταν βγήκε λίγο από το θέμα του πριν, είπε ότι έχουμε την αποπαλλαγή και όσον αφορά την εσωτερική αγορά και την ολοκλήρωσή της. Λοιπόν, πραγματικά δεν βλέπω γιατί δεν πρέπει να συνδυαστεί με αυτό η εκτίμηση επιπτώσεων. Και νωρίτερα όταν εξετάσαμε την έκθεση του ε, το είδαμε. Γιατί λέει ο καθηγητής Μότι ότι εφόσον υπονομεύεται από μια νομοθεσία εσωτερική αγορά, ας πούμε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την ενέργεια και δεν ξέρω τι, και πλήττεται η εσωτερική αγορά, τότε μπορούμε κάλλιστα να ζητήσουμε εκτίμηση επιπτώσεων. Είναι θέμα κοινή λογική. Αυτό που συζητάμε έτσι κι αλλιώς είναι θέμα κοινή λογική. Οπότε, αν προσπαθήσουμε να βάλουμε προτάσει που μιλάνε για εγγύηση και δεν ξέρω τι, για ανεξάρτητος, είναι σαν να πρόκειται για αυτό σκοπό. Όχι. Δεν είναι αυτό που θέλουμε εμεί στη φιλοσοφία μα. Μπορεί να είναι βέβαια λίγο αργά για να αλλάξουμε την έκθεση Νίμπλερ, αλλά αν μη τι άλλο κύριε Βάιλερ, εσείς με... που είσαστε τολμηροί και θαραλέα, μπορείτε να προσπαθήσετε να φροντίσετε έτσι ώστε να βελτιωθεί το τελικό αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ωραία, τελείωσα με την ρητορική μου επιχειρηματολογία, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Βότσον. Να μου πει, συμφωνεί ή όχι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία συνοψίσατε το στόχο μας για το σύστημα εκτιμήσεων επιπτώσεων και το τι θα μας δώσει. Συμφωνώ απόλυτα με την ερμηνεία σας. Και η κυρία Βάιλερ και ο κύριος Κρόιτσμαν έβαλαν το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων σε σημαντικά θέματα εδώ που θέλουμε να τα τονίσουμε γιατί είναι τόσο σημαντικά. Λοιπόν, να αναφερθώ σε αυτά και σε κάποια από αυτά που είπατε εσείς. Για την ανεξαρτησία, αυτό είναι το πιο ευαίσθητο θέμα βέβαια. Ένα από τα θέματα που ίσως δημιουργήσει σύγχυση στη συζήτηση εδώ είναι η σύγκριση με τα εθνικά συστήματα. Ε, όλοι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτές τις συγκρίσεις, γιατί πάντα αντλούνται διδάγματα, πάντοτε εντοπίζονται βέλτιστες πρακτικές, αλλά όλοι μας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες των τεκτενωμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το, η θεσμική δομή των οργάνων μας των τριών κομισιών, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η θεσμική δομή που πρέπει με προσοχή να προστατεύσουμε. Και αν δούμε εθνικές εμπειρίες, η χώρα που μοιάζει πιο πολύ με αυτό που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο εις ό,τι αφορά τη φιλοδοξία για καλύτερη νομοθεσία και εκτίμηση επιπτώσεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν βέβαια διαφορές, ιδιαιτερότητες, αλλά εις ό,τι αφορά την γενικότερη φιλοδοξία μοιάζει πιο πολύ με αυτό που έχουμε εμείς. Τα συστήματα που έχουν στην Ολλανδία και που χαρακτηρίζονται συχνά ανεξάρτητα, στοχεύουν, επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη σημαντική πτυχή της ε, ε, καλύτερης νομοθεσίας που είναι τα διοικητικά βάρη, ο διοικητικός φόρτος και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα ευρύτερο επίπεδο, πιο σύνθετο, πιο πολιτικά ευαίσθητο που μπαίνει στην καρδιά της διαδικασίας διαμόρφωσης και χάραξης πολιτικών. Και αυτό έχουμε υπόψη μας στην προσέγγιση μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το έχουμε, να υπόψη μας όταν κοιτάζουμε τα εθνικά συστήματα. Ε, τώρα, για την ανεξαρτησία πάλι, έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε όταν λέτε ότι η Κομισιόν θέσπισε ένα σύστημα όπου εκείνοι που θα αναπτύσσουν την πολιτική θα είναι οι υπεύθυνοι για να κάνουν και την ανάλυση. Εκείνοι που χαράσουν την πολιτική να καταλαβαίνουν, και αυτό μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουν γιατί κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί κάνουν αυτό που κάνουν με τον τρόπο που το κάνουν, ποιες εναλλακτικέ έχουν και ποια είναι τα ωφέλη και το κόστος των επιλογών τους. Και είναι σημαντικό, όπως είπατε, αυτά τα πρόσωπα που χαράσουν την πολιτική να είναι αυτά που θα κάνουν και τις αναλύσεις. Μετά, ε, μιλήσατε για τον ανεξάρτητο έλεγχο, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα, πολύ ευαίσθητο. Ένα τομέα όπου και η κυρία Νίμπλερ με βάση τη γερμανική εμπειρία έχει διαφορετική προσέγγιση ε, σε σχέση με αυτά που είπαμε εμείς στην Κομισιόν. Ε, εκεί θα θέλαμε πάρα πολύ να δείτε όλοι σας τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο κύριος Μπαρόζο για τον έλεγχο ή τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, όπως τη λέμε. Ε, έχει κάνει ένα συμβούλιο για την εκτίμηση επιπτώσεων από υπαλλήλου ε, της Κομισιόν, ανεξάρτητους από αυτούς που κάνουν την ανάλυση. Και αυτό το Συμβούλιο θα ε, διασφαλίσει την ποιότητα και την αντικειμενικότητα της ανάλυσης και υπάρχουν δυο στοιχεία που θα δούμε εδώ για να διαμορφώσουμε άποψη. Πρώτον, ε, αυτό το Συμβούλιο Εκτίμησης Επιπτώσεων τα τελευταία χρόνια ξαναζήτησε επανάληψη της ανάλυσης γιατί θεώρησε ότι δεν ήταν αρκετά αντικειμενική, σωστή κλπ. Για διάφορους λόγους μπορεί κανείς να ζητήσει επανάληψη της ανάλυσης. Ε, σε 30% των περιπτώσεων έγινε αυτό. Επίσης, οι γνώμες του Συμβουλίου ε, είναι δημοσιευμένοι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευρύτερη επίγνωση των ε, γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο, στους εμπλεκομένους, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της μετέπειτα πολιτικής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Και αν δείτε τις γνωμοδοτήσεις αυτές θα δείτε ότι πολύ συχνά είναι ξεκομμένες, πολύ ομές στη διατύπωσή τους ε, όταν κρίνουν την πρόταση, τις προτάσεις της Κομισιόν και τον αντίκτυπο. Δείτε τα λοιπόν αυτά. Ένα σχετικό θέμα χρειάζεται υπομονή από εσά, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο τώρα εξετάζει τα συστήματα εκτίμησης επιπτώσεων, πώς αξιοποιούνται επίσης από τους επιτρόπους και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ε, περιμένουμε την έκθεση αρχές Σεπτεμβρίου οπότε θα προλάβετε να τη λάβετε υπόψη και στις μελλοντικέ εργασίες και χωρίς να παραβιάσω την εμπιστευτικότητα. Ε, μπορώ να πω ότι θα εντοπίσει όπως όλοι οι καλοί έλεγχοι τα υπέρ και τα κατά, αδυναμίες, δυνατά σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, αλλά αυτό που είναι ενθαρρυντικό στην Κομισιόν είναι ότι επιβεβαιώνει ότι το Συμβούλιο αυτό με τον ανεξάρτητο ελεγκτικό ρόλο που έχει επηρεάζει την ποιότητα της δουλειάς της Κομισιόν, γιατί οδηγεί σε σταδιακές βελτιώσεις που πρέπει να συνεχιστούν στην ποιότητα των αναλύσεών μας και το πιο θεμελιώδες είναι ότι αλλάζει κουλτούρα στην Κομισιόν. Ε, καταλαβαίνουν περισσότερο την ανάγκη να ενσωματώνουν καλύτερη νομοθεσία σε κάθε διαδικασία. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που υποθέτω ότι θα βοηθήσει και το δικό σας έργο μετά τις ε, θερινές διακοπές. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω αναφέρεται στα λεχθέντα από τους, την κυρία Βάιλερ και τον κύριο Κρότσμαν. Η κυρία Βάιλερ ε, μίλησε για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Αυτό διαφοροποιείται από την κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη. Βλέπουμε κοινωνικά ωφέλη, περιβαλλοντικά ωφέλη και κόστη κάθε φορά με ενοποιημένο, ενιαίο, ολοκληρωμένο τρόπο γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι Μόνο όταν τα δούμε όλα αυτά θα μπορέσουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με ένα νόμο και μια νομοθεσία και αν χρειάζεται. Αυτή η ανάλυση θα επηρεάζει επιπτώσεις στους καταναλωτές, στους πολίτες, θα βλέπει να βλέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα αν αυτά εμπλέκονται, θα πρέπει να καλύπτει και όλα αυτά μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Πρέπει να καλύπτει θέματα λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Μόνο αν τα δούμε όλα αυτά μέσα στα πλαίσια μιας ανάλυσης, να δούμε συνέργειες, να δούμε αντισταθμίσματα, αντισταθμίσεις, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε καλή γνώμη για, την, ε, για το νομοθέτημα. Φιλόδοξο το εγχείρημα, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τόσο φιλόδοξα ε, προγράμματα, αλλά ε, έχουν στέρεη βάση, πολιτικά χρειάζονται και επειδή δουλεύουμε και έγκαιρα πιστεύω ότι θα είναι αποτελεσματικά και οι μελέτες εκτιμήσεων επιπτώσεων θα υποβάλλονται έγκαιρα και με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι η γραφειοκρατία και το κόστος ελάχιστα. Αυτά είναι τα βασικά που ήθελα να πω σήμερα. Προφανώς είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία θα θελήσετε σε οποιοδήποτε στάδιο των διαβουλεύσεών σας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Την Κομισιόν, ε, πολύ σαφής η τοποθέτηση. Έχω την ε, Έχω διαβάσει την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αν και ως πρόεδρος κανονικά δεν πρέπει να πω τίποτα, γιατί το ελεγκτικό συνεδρίο ε, συμμετείχε σε μία συζήτηση όπου αναλύσαμε λιγάκι την σημασία των μελετών ε, επιπτώσεων, ας πούμε, ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ήταν σημαντική, εν η έκθεση αυτή. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Κυρία Βάιλε, θέλετε να συνοψίσετε να μιλήσετε επίσης και για το χρονοδιάγραμμα, το οποίο φυσικά συνδέεται και με τις προθέσεις κυρίας Νίμπλερ, που είναι η εξουσίας αρμόδια συντάκτρια. Να, να πω και κάτι τώρα στο τέλος. Καταρχήν πρόσεξα, κύριε Πρόεδρε, ότι δώσατε στην ομάδα ECR πολύ χρόνο. Παρά είσαστε γενναιόδωρος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ε, Προς τον κύριο Κρόιτσμα να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Το θέμα επικουρικότητα, όπως το ερμηνεύσατε, δεν είναι όπως το εννοεί η κυρία Νίμπλερ. Η εναλλακτική, δημόσιο ή ιδιωτικό, είναι ένα θέμα. Αλλά ε, όπως θέλει να κάνει τον έλεγχο επικουρικότητας, είναι αν θα πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη ή αν θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Το πανάρχιο, το παμπάλαιο ερώτημα που γίνεται ακόμα πιο έντονο μετά τη Λισαβόνα και που καμιά φορά έχουμε διαφορετική άποψη εμείς από τους εθνικούς βουλευτές. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα κοιτάξουμε. Κύριε Πρόεδρε, για τις εκπρόθεσμες ή καθυστερούμενες πληρωμές, late payments, πολύ σωστά το είπατε και το αναφέρατε. Είναι πολύ χρήσιμη η μελέτη εκτίμηση επιπτώσεων σε αυτά τα θέματα και οι μόνοι που έκαναν κριτική δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι, οι stakeholders όπως λέμε, δεν ήταν ο κλάδος, η βιομηχανία, δεν ήταν οι διοικήσεις, ήταν παραδόξως κάποια κράτη-μέλη που δεν τους άρεσαν ορισμένα νούμερα. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό στην πράξη. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε οι σκιώδη της ομάδας ECR ή όπως και να είστε, ότι η ανάθεση σε εξωτερικούς προφανώς δεν εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Όχι, ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Οπότε αν μιλήσουμε για ανεξάρτητη γνωμοδότηση, δεν επιτρέπεται να το κάνει η Κομισιόν. Αυτό είναι λάθος και στερείται οποιασδήποτε λογικής βάσης και προσκρούει στην εμπειρία μας. Το independent σημαίνει άλλο πράγμα για μένα. Ξέρω περιπτώσεις όπου η Price Waterhouse ή ε, κάποια άλλη ανέλαβε να κάνει μια έρευνα για την δημοσιονομική ρύθμιση και για ε, δημοσιονομικούς ε, κανόνες και νομοθεσίες και εκεί αμφισβητείται η ανεξαρτησία τους. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ξέρω τη δουλειά της Κομισιόν και πριν από την εκτίμηση για τις ε, εκπρόθεσμες πληρωμές και είμαι πεπισμένη. Δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια και πιο σωστά πολιτικά από ότι σε εθνικό επίπεδο. Εάν συνέβαινε αυτό και αν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, δεν θα συζητούσαμε σήμερα. Ούτε θα συζητούσαμε θέματα όπως για παράδειγμα ε, πτώσεις στους καταναλωτές που θέλουμε να τα δούμε καλύτερα γιατί μέχρι τώρα δεν τα είχαμε δει καλά όπως έπρεπε και κάποια άλλα πράγματα που χρειάζονται διορθώσεις. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα έχω μια παράκληση. Αν αληθεύει ότι η Κομισιόν στις θερινές διακοπές θα επεξεργαστεί πολλά έγγραφα τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να τα έχουμε. Θα μας έρθουν γύρω στις 31 Αυγούστου, τέλος πάντων κάπου στα τέλη Αυγούστου. Παρακαλώ να γίνει ξανά μια ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή, αφού, αφού λάβουμε τα έγγραφα από την Κομισιόν και, με συμμετοχή, και να κάνουμε και μια ακρόαση όχι να, η Επιτροπή να το κάνει, ίσως να συμμετάσχουμε σε μια ακρόαση της Νομικής Επιτροπής. Γιατί κάτι θα κάνουν. Ίσως θα φωνάξουν και εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, ίσως και κάποιον Αμερικανό καλό είναι να πάμε και να συμμετάσχουμε εμείς, όχι να το κάνουμε εμείς να το οργανώσουμε, αλλά να συμμετέχουμε σε αυτά που θα κάνει η Νομική Επιτροπή, σε στενή συνεργασία, γιατί αυτό θα βοηθήσει. Και πριν υποβάλω την έκθεσή μου, θα ήθελα να κάνουμε πάλι μια ανταλλαγή απόψεων. Και ίσως να καταγράψω ορισμένα θέματα, να τα έχουμε γραπτός. Γίνεται και αυτό. Και πρέπει να κινηθούμε έγκαιρα πριν από την ψηφοφορία στην Νομική Επιτροπή, γιατί μας ενδιαφέρει τα δικά μας τα θέματα, η δική μας ε, προβληματική να ληφθεί υπόψη από την Νομική Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Βάιλερ για αυτά που είπατε. Μιλάτε ουσιαστικά για την έκθεση της, ε, του Ελληνικού Συνεδρίου για τις, τα κείμενα και τις μελέτες ε, αντικτύπου. Ε, το τεχνικό συνόριο μπορεί να έρθει και να παρουσιάσει την έκθεση στο Κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να το δείτε με την κυρία Νίμπλερ. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνετε. Εγώ πήρα ένα αντίτυπο, είχα αυτό το προνόμιο, αλλά καλό είναι να το δείτε κι εσείς. Επίσης μια κοινή ακρόαση, καλό θα ήταν. Ε, με την, μαζί με την νομική επιτροπή, του ή όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου είναι προσκεκλημένα. Ε, ακόμα και προσκεκλημένοι από τον άλλο νομοθετικό βραχίωνα. Μπορείτε να το συζητήσετε με την κυρία Νίμπλερ για να το κάνετε. Σε ό,τι αφορά το χρόνο μιλίας. είναι το τελευταίο σημείο. Δεν ήξερα ότι, δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε περιορισμένο χρόνο. Ξέρω βεβαίω ότι ήμουν γενναιόδωρος και με την ομάδα μου αλλά και με τον εαυτό μου. Ε, είναι ένα από τα πάθη μου αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Βάιλερ, περιμένουμε την εκθεσή σας μετά τις διακοπές και μέχρι τότε ελπίζω ε, να έχετε ολοκληρώσει και την, το κείμενο για τις καθυστερημένες πληρωμές. Ε, είσαστε από τους πιο σκληρά εργαζόμενους βουλευτές αυτής της Επιτροπής. Αυτά. Κλείνουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Θα συνεδριάσουμε ξανά Δευτέρα, 13 Ιουλίου, όχι 12 Ιουλίου, 3 η ώρα το απόγευμα και εν συνεχεία, α, σε αυτή την αίθουσα, έτσι, σε αυτή την αίθουσα και επίσης την Τρίτη, 13 Ιουλίου από τις 9 μέχρι το 10.30 και συμφωνήσαμε στους συντονιστές να γίνει μια σύντομη συνεδρίαση το απόγευμα, 3 με 5 στις 13 Ιουλίου. Εντάξει, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Τελείωσε η συνεδρίαση.